Αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ήρθατε. Καλωσορίζω και τον Ρουμανό Υπουργό Οικονομικών, το Αίγιον Ορλάντο Τεοντορόβιτσι. Καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε που ήρθατε. Πριν αρχίσουμε τον οικονομικό διάλογο με τον πρόεδρο του ΕΚΟΦΗΝ, να κρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Παρατηρήσεις, όχι. Ωραία. Ανακοινώσει του Πρόεδρου αύριο θα γίνουν πριν την ψηφοφορία. Οπότε περνάμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης που είναι οικονομικός διάλογος με τον πρόεδρο του ΕΚΟΦΗΝ, τον κύριο Έγγεν Ορλάντο Τεοδωρόβιτσι. Καλώς ήρθατε. Συγχαρητήρια και ό,τι καλύτερο εύχομαι για το εξάμεινο αυτό της Προεδρίας σας. Εμείς προσβλέπουμε σε συνεργασία με την Ρουμανική Προεδρία με ένα θετικό, καλό κλίμα για να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατόν αποτελέσματα. Σήμερα ο κύριος Τεοντορότσι θα μας παρουσιάσει τις προτεραιότητες της Ρουμανικής Προεδρίας. Καλωσορίζουμε το πρόγραμμα της Ρουμανικής Προεδρίας και σας ευχαριστούμε για όσα θέλετε για την σύγκληση, σύγκληση προς τα πάνω βέβαια, ανάπτυξη, επενδύσεις, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, κοινωνική, δαφική συνοχή, οικονομική συνοχή, δικαιοσύνη και ενίσχυση του κοινωνικού πυλώνα. Αύριο θα συνεδριάσει για πρώτη φορά το ΕΚΟΦΗΝ υπό τη δικιά σας προεδρία. Εκεί θα συζητήσετε διάφορους φακέλους που είναι πολύ σημαντικοί και διασφαλίζουν τη σύγκληση βάσει της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ευρώπη. Εδώ θέλω να τονίσω όλος ιδιαίτερος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δώσει εντολές διαπραγμάτευσης και για το InvestEU και για την μεταρρύθμιση του ΕΦΣΥ, οπότε σας ζητούμε από εσάς και από το Συμβούλιο να προχωρήσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα για να μπορέσουμε να υιοθετήσουμε και συμφωνία για την ενίσχυση των επενδύσεων. Το Κοινοβούλιο και οι βουλευτές έχουν στείλει επιστολή ζητούντας ε, διαπραγματευτική εντολή για ολόκληρο το φάκελο των μεταρρυθμίσεων ΕΦΣΑ. Οπότε ελπίζω αυτό να το πετύχουμε εμβάθυνση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, φορολογία, είναι και αυτοί οι τομεί που θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Όπως επίσης θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και στους τριμερείς διαλόγους και σε 9 ή 10 θέματα ε, για τα οποία έχουμε ήδη ξεκινήσει τις συζητήσεις με την Προεδρία σας. Θα συνεχίσουμε. Έχουμε ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο πρόγραμμα και πάλι σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να πετύχει η Προεδρία σας. Ευχαριστούμε πολύ και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές. Πρώτα απ' όλα, σας εύχομαι καλή χρονιά. Με κάθε επιτυχία, υγεία και να ξέρετε ότι είναι μεγάλη τιμή για μένα που βρίσκομαι εδώ μαζί σας για αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων με την Ρουμανική Προεδρία ε, στα πλαίσια της Οικονομικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και έτσι θα μπορέσουμε να ανταλλάξουμε απόψεις, να σας ενημερώσω για τους στόχους μας και τις ε, ελπίδες μας για το επόμενο εξάμεινο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους Ευρωβουλευτές για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα. Ευχαριστώ και την προηγούμενη Προεδρία αλλά και της ε, Βουλγαρίας, ε, της Αυστρίας, των προηγούμενων Προεδριών που επίσης βοήθησαν πολύ. Ποιοι είναι οι βασικοί πυλώνες της ε, Προεδρίας μας, θα σας πω και ποια είναι η κατάσταση οικονομική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης θα σας πω και ποια είναι τα σχέδια της Ρουμανικής Προεδρίας στα θέματα τα οικονομικά, νομισματικά και φορολογίας και μετά θα απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν διάφορες επιθυμίες και ανησυχίες, κάτι το οποίο βρίσκεται στην καρδιά ε, της Ρουμανικής Προεδρίας και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η φιλοδοξία μας είναι να προχωρήσουμε και να ε, κλείσουμε ε, διάφορα νομοθετικά ζητήματα όσο γίνεται πιο γρήγορα. Η Ρουμανική Προεδρία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου σε μια πολύ σημαντική στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση όπου έχουμε πάρα πολλές προκλήσεις. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν πρέπει να διατηρηθεί η ακαιρεότητα του ευρωπαϊκού σχεδίου και η συνοχή μεταξύ των χωρών μελών. Αυτή είναι η βασική στόχη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι κάτι το, στο οποίο θέλουμε και εμείς να συνεισφέρουμε. Όμως είμαστε ρεαλιστές συγχρόνως, αλλά και φιλόδοξοι. Γνωρίζουμε ότι η Προεδρία αυτή έρχεται στο τέλος ε, της θητείας και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε από κοινού προσπάθεια και να δείξουμε ισχυρή βούληση τόσο το Συμβούλιο όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και είμαι σίγουρος ότι όλοι θα είμαστε αποτελεσματικοί και θα έχουμε μεγάλη πρόοδο σε πολλούς και διαφορετικούς φακέλους. Τώρα ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ την ε, ε, Ρουμανική Προεδρία είναι ο εντοπισμός ευκαιριών και η δημιουργία ευκαιριών για τους Ευρωπαίους πολίτες. Είχαμε τα 100 χρόνια ε, της Ένωσής μας πέρυσι στη Ρουμανία. Πάνω από 50 χρόνια δημοκρατίας κράτους δικαίου και μπήκαμε και στον ελεύθερο κόσμο, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την Ευρώπη. Πριν από 30 χρόνια το όνειρο αυτό φαινόταν σαν κάτι το αδύνατο για μας. Τώρα, μάλλον τότε, ε, στην Ευρώπη φτάναμε μόνο μέσα από κάποια μουσική, μέσα από κάποια παράνομα, κάποιους παράνομους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Προσπαθούμε όμως σήμερα να χτίσουμε όλα αυτά τα οποία στερηθήκαμε όλα τα χρόνια που δεν είχαμε πρόσβαση στην Ευρώπη. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά που βρίσκομαι και τι σημαίνει η στήριξη του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του κ. Ταγιάννη, που στις 10 Ιανουαρίου μίλησε για την Ρουμανική Προεδρία. Μίλησε για τη σύγκληση που είναι πράγματι μια ευρωπαϊκή αξία. Εμείς πιστεύουμε ότι διαφορές ε, μπορεί να υπάρχουν, αλλά το να μας χωρίζουν αυτό δεν είναι ευρωπαϊκή αξία. Γι' αυτό λοιπόν η Ρουμανική Προεδρία θα είναι υπέρ της σύγκλησης στην Ευρώπη. Η βασική στόχη μας λοιπόν θα είναι ακριβώς αυτό, η σύγκληση στην Ευρώπη. Τώρα όσον αφορά ε, την ίση μεταχείριση μεταξύ χωρών μελών και μεταξύ πολιτών, η Ρουμανία θα δραστηριοποιηθεί προκειμένου να παγιωθεί η ευρωπαϊκή διαδικασία και να πετύχουμε πρόοδο στον δημοσιονομικό τομέα και τον δημοσιονομικό και το φορολογικό και τον οικονομικό και να στηρίξουμε οικονομικές μεταρρυθμίσεις προ όφελο των χωρών μελών και των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει περισσότερη δύναμη, να ευημερεί περισσότερο, ώστε να μπορέσουν εξίσου όλοι οι πολίτες να υποφεληθούν από την ασφάλεια, ε, την ευημερία, και να έχουν δυνατότητες ανάπτυξης. Εμείς θέλουμε να διασφαλίσουμε μια ευρωπαϊκή προεδρία με ανάπτυξη για την Ευρώπη, ξέροντας ότι τώρα έχουμε μεσαία επίπεδα. Ε, η πρόγνωση που έχουμε είναι αρκετά αισιόδοξη σήμερα, παρόλο που σίγουρα θα υπάρξει κάποια επιβράδυνση στους ε, ρυθμούς. Υπάρχουν κίνδυνοι, υπάρχουν εντάσεις στο εμπόριο, σε διάφορες πολιτικές που ακολουθούμε, υπάρχουν γεωπολιτικά προβλήματα, υπάρχει ρευστότητα στις οικονομικές αγορές και γι' αυτό εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούμε να καθίσουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Αντίθετα, πρέπει να υποφεληθούμε από την θετική ευκαιρία, ε, συγκυρία που έχουμε για να ενισχύσουμε τη θέση μας ακόμα περισσότερο. Θέλουμε διαφάνεια και θέλουμε να συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή όλες οι χώρες μέλη και όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα επίσης όρις. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά έχοντας υπάρξει βουλευτή στο Ρουμανικό Κοινοβούλιο τι σημαίνει η συνεργασία μεταξύ μας. Πώς θα μπορέσει να υπάρξει καλή συνεργασία ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Για μας είναι ζωτική σημασίας. Διότι έχουμε πολλούς τριμερείς διαλόγους και συζητήσεις μεταξύ μας, συνδιαλλαγή πριν από τις επόμενες ευρωεκλογέ. Στους έξι αυτούς μήνες λοιπόν θα δουλέψουμε για την σύγκληση στο ΕΚΟΦΗΝ και στόχος μας είναι να προωθήσουμε την οικονομική και την κοινωνική σύγκληση και να βελτιώσουμε τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Θα επικεντρωθούμε στη μείωση των διαφορών στην ανάπτυξη που υπάρχουν μεταξύ περιφερειών και μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών και οικονομικών κατηγοριών για να ενισχύσουμε τη συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν θέλουμε να επικεντρωθούμε στα εξή. Πρώτον, θέλουμε να εμβαθύνουμε περισσότερο στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση να υπάρξει παγίωση της Τραπεζικής Ένωσης και παρετέρω ανάπτυξη της Ένωσης Κεφαλαιογορών. Θέλουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και να υπάρχει και σωστός συντονισμός και συνεργασία στις οικονομικές πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας και να ενισχύσουμε την ατοχή μας. Η Ρουμανική Προεδρία αναγνωρίζει ότι η, Ευρωπαϊκή, Οικονομική και Νομισματική Ένωση πρέπει να ολοκληρωθεί και ότι αυτό υπάρχει στο χάρτη πορείας που είχαμε και θα τονίσουμε επίσης και τώρα το Μάρτιο του 2019. Σας ευχαριστώ για τις δικές σας προσπάθειες προκειμένου να βαθύνουμε περισσότερο στην ΟΝΕ. Η Ευρώπη κατάφερε να ανακάμψει από την ε, κρίση σε έναν μεγάλο βαθμό. Η Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική σήμερα είναι ιδιαίτερα ισχυρή, αλλά πρέπει να κάνουμε και άλλες προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ότι θα μπορέσουμε να κινηθούμε με το πλήρες δυναμικό μας για να πετύχουμε την ευημερία και τη σταθερότητα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διάσκεψη κορυφής του Δεκεμβρίου του 2018 έθεσε ε, του, της βάσης για να βαθύνουμε περισσότερο στην ΟΝΕ. Συμφωνήθηκε να αλλάξουμε την συνθήκη και μέσα στο 2019 θα προετοιμαστούμε γι' αυτό. Πρέπει να υπάρξει πρόοδος όσον αφορά την Τραπεζική Ένωση και την Ένωση Κεφαλαγορών. Τον Ιούνιο του 2019 θα πρέπει να έχουμε κάποια συμπεράσματα. Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά τώρα ε, του προπολογισμού για τη σύγκληση στην Ευρωζώνη. Και εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την οικονομική πραγματικότητα που ισχύει στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τα βήματα που θέλουμε να αναλάβουμε τώρα, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι λειτουργούμε με μια ανοιχτή διαδικασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να συμμετέχουν δηλαδή και οι χώρες οι οποίες δεν είναι μέλη στην Ευρωζώνη. Χρειάζεται ένα στέρεο οικονομικό τομέα, κάτι από το οποίο έχουν αποφεληθούν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτε. Γι' αυτό και πρέπει να κάνουμε μεγάλη πρόοδο για την Τραπεζική Ένωση. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ του προκατόχου μα στην Αυστριακή Προεδρία, αλλά βέβαια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πολιτική συμφωνία στην οποία κατέληξαν στο τραπεζικό πακέτο. Για την εφαρμογή του θα αναλυθούν παρετέρω μέτρα για τη μείωση των κινδύνων. Προς το παρόν δουλεύουμε εντατικά για να ολοκληρωθεί το πακέτο και ελπίζουμε ότι θα υιοθετηθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα. Χρειάζεται επίσης και ένα κοινό backstop, ένα δίκτυο ασφαλείας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Τραπεζική Ένωση. Και η διάσκεψη του Δεκεμβρίου ακριβώς έθεσε τους όρους αναφοράς για το δίκτυο αυτό ασφάλειας, για αυτό το backstop πώς δηλαδή θα λειτουργήσει αυτό. Φυσικά χρειάζεται συντονισμός με την Προεδρία του Eurogroup και πρέπει να δουλέψουμε και για άλλα θέματα τα οποία μπαίνουν στη μέση, όπως η εμβάθυνση στην ΟΝΕ. Τέλος, αλλά όχι και λιγότερο σημαντικό, όσον αφορά τις προτεραιότητες της Τραπεζικής Ένωσης. Εδώ μιλάμε για νομοθετικές προτάσεις, οι οποίες θα προσπαθήσουν να μειώσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τον όγκο του. Δεν θέλουμε να συσσωρεύσουμε και πάλι τέτοια μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Και είναι πολύ καλή η συμφωνία που πετύχαμε τον Ιούλιο για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Και όσον αφορά την οδηγία για το MPL, ελπίζουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα να πετύχουμε συμφωνία για τις ε, διαπραγματευτικές θέσεις στο Συμβούλιο για τις δευτερεύουσες αγορές. Έρχομαι τώρα στους ε, φραγμούς, εμπόδια που έχουμε για την ε, Ένωση Κεφαλαιογορών. Εδώ πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο πάνω σε νομοθετική πρόταση για να μειωθούν οι διαφορές μεταξύ των διάφορων δικαιοδοσιών και να υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες για τους επενδυτές και πρόσβαση σε όσο γίνεται μεγαλύτερο εύρος οικονομικών πόρων. Δουλεύουμε πολύ σκληρά, λοιπόν, και θα συνεχίσουμε τους ε, επόμενους μήνες. Και θα έρχομαι στα, στους 7 φακέλους πάνω στους οποίους ήδη δουλεύουμε και θα έχουμε διάλογο. Πρώτα απ' όλα υπάρχει το πακέτο βιώσιμων οικονομικών. Η πρόταση είναι πολύ σημαντική για να πετύχουμε ε, κλιματικούς στόχους, περιβαλλοντικούς στόχους, κοινωνικούς ενεργειακούς ε, στόχους σύμφωνα με τη Συμφωνία των Παρισίων του 2016 και την ε, ατζέντα για την βιώσιμη ανάπτυξη του ΟΗΕ ενώπιση του 2030. Εργαζόμαστε λοιπόν για τους τριμερείς διαλόγους ε, που θα έχουμε σύντομα και θα είμαστε σε στενή επαφή μαζί σας για να τηρείτε ο κανόνας της διαφάνειας. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα για την ΟΝΕ είναι η κατανομή πόρων διασυνοριακά. Και αυτό είναι ένα σημαντικό πακέτο για να μειωθούν τα εμπόδια που υπάρχουν σήμερα, να μειωθεί επίσης και το κόστος, αλλά να ενισχύσουμε και την ανταγωνιστικότητα και τη δυνατότητα οι καταναλωτές να έχουν περισσότερες ε, εναλλακτικέ και επιλογές. Ελπίζουμε να ολοκληρώσουμε πριν το τέλος της θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ερχόμαστε τώρα στα εγγυημένα ομόλογα. Εδώ θα συνεισφέρει το θέμα αυτό στην διεύρυνση των κεφαλαϊκών αγορών. Αυτές οι νομοθετικές πράξεις θα βελτιώσουν την ασφάλεια για τον επενδυτή και θα δώσει δυνατότητες για αγορές οι οποίες είναι λιγότερο αναπτυγμένες. Έχουμε ήδη ένα πρώτο τριμερή διάλογο και ελπίζουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα να καταλήξουμε σε συμφωνία μαζί σας ε, για το πακέτο αυτό όσον αφορά τα εγκυμένα ομόλογα. Έπειτα έχουμε τα εποπτικά μέτρα <clears throat> για τους επενδυτές. <clears throat> Εδώ υπάρχουν απαιτήσει εποπτικές και για το θέμα αυτό έχουμε προχωρήσει σε διατάξεις βάσει διάφορων business model και ε, προφίλα κινδύνου ώστε να μην πληγεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των ε, τραπεζών. Χρειαζόμαστε εντολή βέβαια διαπραγματευτική για το πακέτο αυτό και τώρα περιμένουμε να αρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις μαζί σας ήδη από αυτή τη βδομάδα. Ένα άλλο θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό έχει να κάνει με τους κεντρικούς ομολόγους και την σχετική εποπτεία, το ΕΜΥΡ. Η πρόταση αυτή με τις τροπολογίες ε, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα συνεισφέρει στην ενίσχυση του εποπτικού συστήματος τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στους τρίτους ε, κεντρικούς ε, ομολόγους σε τρίτες χώρες. Έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη μας την πολυπλοκότητα που έχει το θέμα των αποζημιώσεων. Ο πρώτος τριμερής διάλογος έλαβε ήδη χώρα την προηγούμενη εβδομάδα και ελπίζουμε ότι θα καταλήξουμε σε πολιτική συμφωνία μαζί σας όσο γίνεται πιο γρήγορα. Επίσης είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε και όσον αφορά την αναθεώρηση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών. Ήδη στις 19 Δεκεμβρίου του 2018 η Κοροπέρ υιοθέτησε διαπραγματευτική εντολή όσον αφορά το θέμα της ε, αντιμετώπισης της ε, νομιμοποίησης παράνομου χρήματος. Προχωρούμε λοιπόν, αλλά πιστεύουμε ότι οι τροπολογίες επίγουν, ιδίως όσον αφορά ε, το πλαίσιο πρόσφατων υποθέσεων που είχαμε με προσπάθειες νομιμοποίησης παράνομου χρήματος. Αύριο το Συμβούλιο θα συζητήσει τα επόμενα βήματα για το φάκελο αυτό και θα σας ενημερώσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Επιπλέον, έχουμε και ε, το τεχνικό σκέλος του κανονισμού εμίρ Ρεφίτ για τις υποδομές της ευρωπαϊκής αγοράς. Ελπίζουμε ότι εδώ θα προχωρήσουμε γρήγορα και είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε γρήγορα και για άλλες προτάσεις για το FinTech πρόγραμμα δράσης ή το crowdfunding. Ελπίζουμε ότι θα πετύχουμε πρόοδο σύντομα για να πετύχουμε και τους στόχους μας, αλλά γι' αυτό χρειαζόμαστε και τη δική σας στήριξη. Έτσι θα μπορέσουμε μαζί να πετύχουμε πρόοδο σε πολλούς φακέλους μέσα στο λίγο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας μέχρι τις ευρωεκλογές. Τώρα έρχομαι σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τις προσδοκίες των ε, πολιτών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η δίκαια φορολόγηση. Εδώ θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για δίκαια φορολογικά συστήματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τις επιχειρήσεις και για τις φορολογικές αρχές. Επίσης θα δουλέψουμε εντατικά και για την υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά πληρωμές που γίνονται από τη συλλογή ε, ΦΠΑ, φόρου προστιθέμενης αξίας. Πριν όμως υιοθετήσουμε μέτρα για ένα οριστικό σύστημα, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν δημιουργούμε νέες ευκαιρίες για απάτες στον τομέα του ΦΠΑ. Και αυτό, η προσπάθεια αυτή έχει ήδη ξεκινήσει. Κάποιες αλλαγές θα πρέπει να γίνουν για να υπάρξει βελτίωση στην συνεργασία μεταξύ των διοικητικών αρχών των χωρών μελών. Το Συμβούλιο θα συμφωνήσει για ένα νέο κανονισμό όσον αφορά τον ΦΠΑ για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα απάτης, να τα αποφεύγουμε. Θέλουμε τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο γίνεται πιο γρήγορα για το ΦΠΑ. Όπω γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα υιοθέτησε μία ανακοίνωση για την ψηφοφορία με ενισχυμένη ψηφοφορία και για τι νομοθετικέ διαδικασίε στον τομέα τη φορολόγηση. Υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ με την αποτελεσματικότητά μα Όταν εγκρίνουμε φορολογικά μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε θέλουμε και τη δικιά σας άποψη για το θέμα αυτό και οποιοδήποτε πρωτοβουλία παίρνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, προηγουμένως πρέπει βεβαίως να έχει αξιολογηθεί και εκτιμηθεί και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το στάδιο Πάντως θέλω να σας πω ότι εγώ θα το θέσω το ζήτημα για συζήτηση στα πλαίσια του ΕΚΟΦΗΝ και είμαι σίγουρος ότι όλοι μαζί θα πετύχουμε μία λύση για το πώς μπορεί να εφαρμοστεί η ιδέα αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ποια θα πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις αν ακολουθήσουμε αυτή την πορεία. Συγχρόνως πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια το Συμβούλιο έχει νομοθετήσει πολύ γρήγορα. Παρά την απέτηση για ομοφωνία που υπάρχει τώρα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν το έργο μας και όσον αφορά την οδηγία για τις ψηφιακές υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με τη φορολογία. Θέλουμε μια κοινή προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την φορολόγηση αυτή της ψηφιακής οικονομίας. Συγγνώμη, πρόκειται για την ε, ψηφιακή οικονομία και την φορολόγησή της. Πρέπει να υπάρχει μια ενιαία προσέγγιση για τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΣΑ η Προεδρία θα στηρίξει μια επικοδομητική συζήτηση επίσης για την κοινή φορολογική βάση και θα συνεχίσει το έργο για τα τεχνικά στοιχεία. Και θα βασιστούμε φυσικά στην καλή δουλειά που έχει ήδη γίνει από τις προηγούμενες Προεδρίες. Θα ολοκληρώσουμε επίσης τον κανονισμό φυσκάλης μετά το 2020. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα συνεργασίας, ώστε οι εθνικές φορολογικές αρχές να έχουν ένα σύστημα ανταλλαγής και να βελτιώσουν την πραγματογνωμοσύνη τους. Η Προεδρία μας επίσης καλωσορίζει την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτό το ζήτημα και προσβλέπουμε σε μια γρήγορη πολιτική συμφωνία. Τώρα όσον αφορά τη φορολογική διαφάνεια και τον φορολογικό ανταγωνισμό, θα δουλέψουμε μαζί σε διακυβερνητικό επίπεδο για τον συντονισμό των φορολογικών θεμάτων. Θα υπάρχει ένας κατάλογος με μη συνεργαζόμενες φορολογικές δικαιοδοσίες βάσει των υποχρεώσεων που θα αναλάβουν τρίτες χώρες. Και η δέσμευση αυτή λήφθη στα τέλη του 2018. Το ΕΚΟΦΗΝ και η Ρουμανική Προεδρία ετοιμάζει ένα τέτοιο κατάλογο με συνεργαζόμενο δικαιοδοσών. Όσον αφορά τώρα τους φόρους πολυτελείας, η Ρουμανική Προεδρία θέλει να συντάξει μια οδηγία με ένα ειδικό καθεστώς για τους φόρους πολυτελείας που θα προσφέρουν ένα σαφές νομικό πλαίσιο και θα οδηγήσει ε, σε μια σταθερότητα στην αγορά και θα αποφεύγεται η φοροδιαφυγή. Θέλουμε και εδώ την συνεργασία σας και για την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων τώρα. Η Ρουμανική Προεδρία θέλει να ολοκληρωθεί η ρύθμιση για τη χρηματοδότηση των εξωτερικών συνόρων. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει πρόοδος επίσης και η τα όσον αφορά το σχετικό κανονισμό για μετά το 2020. Στηρίζουμε τις διαδικασίες για ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Τελωνίων. Χρειαζόμαστε τη συνεργασία βέβαια και των τελωνιακών αρχών. Τέλος, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι κάτι πολύ σημαντικό για το συντονισμό της ε, οικονομικής μας ε, πολιτικής και είμαστε ικανοποιημένοι από την ε, έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την, την επισκόπηση για την ετήσια ανάπτυξη που θέτει πολιτικέ προτεραιότητε, που είναι η απασχόληση και η ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες μέλη ξεκινώντα από το 2019, από το εξάμενο δηλαδή του 2019 που θα περιλαμβάνει αυτά τα στοιχεία. Ενθαρρύνουμε για την εφαρμογή επίση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων. Σαν πρώτο βήμα, εμείς προτείνουμε να υπάρξει πρόοδος στο πρόγραμμα Invest EU καταρχήν και μετά θέλουμε να δούμε αν θα πετύχουμε και συνένεση για το πρόγραμμα στήριξης των μεταρρυθμίσεων. Πιστεύουμε ότι μπορεί να συνεισφέρει στην όθηση για παρετέρω ανάπτυξη. Η πρώτη συζήτηση με τους Υπουργούς Οικονομικών για το Invest EU θα λάβει χώρα αύριο, να ξέρετε, στην πρώτη συνάντηση ΕΚΟΦΗΝ. Εκεί θα πιστήσω την προσοχή των συναδέρφων σε διάφορα σημαντικά θέματα που έχουν να κάνουν με το προσανατολισμό των διαπραγματεύσεων για αυτό το θέμα. Είναι επίση ζωτική σημασία να εντοπίσουμε διάφορες λύσεις για το πρόγραμμα Invest EU. Και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μία δίκαια γεωγραφική κατανομή για τους ευρωπαϊκούς σπόρους τα ευρωπαϊκά κονδύλια και να ενισχύσουμε τη δυνατότητα απορρόφησης των χωρών μελών για όλα τα προγράμματα. Η Ρωμανική Προεδρία θα διασφαλίσει ότι θα έχουμε και απαλληλογή για τον προβλησμό το 2017 και θα ξεκινήσουμε και με τον προπολισμό του 2020. Επίσης θέλω να σημειώσω και κάτι πολύ σημαντικό για μα. Το πρώτο πλεονέκτημα του να είναι κανεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τα κονδύλια που παίρνει κάθε χώρα, είναι για τις αρχές και τις αξίες που συνοδεύουν την προσχώρηση της κάθε χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι το πολύτιμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι που μας κάνει διαφορετικούς καλύτερους και περισσότερο αντοχής. Είμαι αποφασισμένος και είμαι σίγουρος ότι μόνο ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα, πολύ περισσότερα από ό,τι θα κάναμε μόνοι μας. Στη Ρουμανία 24 Ιανουαρίου γιορτάζουμε την ενοποίηση των Ρουμανικών Πρικυπάτων το 1850. Τότε ήταν που δημιουργήσαμε την πρώτη ένωση και οι βάσεις γράφτηκαν από επαναστάτες. Τα λόγια που αναφέρονται εκεί είναι ότι μαζί θα γίνουμε περισσότερο ισχυροί. Και αυτό ακριβώς είναι και το έμβλημά μας. Και δεν πρόκειται μόνο για τους Ρουμάνους, πρόκειται για όλα τα έθνη. Σεβόμαστε τη γλώσσα που μιλάμε, ε, το πώς γράφουμε. Έτσι μόνο θα είμαστε περισσότερο ισχυροί μαζί. Είμαι αποφασισμένος λοιπόν. Τα αποτελέσματα για αποτελέσματα από τη Ρουμανική Προεδρία. Ελπίζουμε σε επιτυχίες και όλα αυτά θα είναι μια κοινή επιτυχία όλων μας μαζί και θα τα καταφέρουμε καλύτερα αν δεν ξεχνάμε αυτό που είπε ένας από τους ιδρυτές πατέρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ζαμονέ, ο οποίος είπε αυτό που είναι σημαντικό δεν είναι μόνο να είναι κανείς αισιόδοξο ή απεσιόδοξο, αλλά να είναι αποφασισμένος να πετύχει. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank Σε ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Υπουργέ για την συνολική σας αυτή παρουσίαση. Ας ξεκινήσουμε τώρα με τις παρεμβάσεις των βουλευτών. Ο κύριος Μουρεσάν πρώτος για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σας εύχομαι καλή πτυχία το επόμενο εξάμεινο. Έχω δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα μιλήστε για την Οικονομική και την Νομισματική Ένωση και την διαδικασία αυτή που βρίσκεται εν εξελίξη. Η Κομισιόν το τέλος του 2017 είχε πει ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό νομισματικό ταμείο και στο τέλος του 2018 μίλησε για έναν επενδυτικό μηχανισμό. Εγώ όταν το άκουσα υποστήριξα την ιδέα και είπα ότι θα πρέπει να περιλάβει και χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωζώνης. Σας ερωτώ λοιπόν τι θα κάνετε συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της ε, Προεδρίας σας έτσι ώστε τα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία δεν είναι με ακόμα μέλη της Ευρωζώνης να περιληφθούν θεωρείτε ότι θα συμμετάσχουν τελικά σε αυτά τα δύο έργα. Μετά, για τις χώρες ε, που δεν είναι μέλη της Ευρωζώνης, πώς θα μπορέσουν ακριβώς να ωφεληθούν από αυτά τα δύο έργα. Και αν βλέπετε κάποια διαφορά μεταξύ των κρατών εκείνων που είναι μέλη του συναλλαγματικού μηχανισμού, ε, του δεύτερου μηχανισμού συναλλαγματικών συντομιών και όσων δεν είναι. Δεύτερον. Έχουμε το πρόγραμμα εργασίας της ε, Ρουμανικής ε, Προεδρίας. Εκεί πέρα υπάρχει ένας, ε, ένα θέμα το οποίο θα περιλάβει εμάς ως Κοινοβούλιο και εσάς ως Συμβούλιο και αφορά τους ειδικού φόρους κατανάλωσης και την πρόταση της Κομισιόν. Αυτό είναι το μόνο το οποίο απομένει να ολοκληρωθεί στα έγγραφα του ΕΚΟΦΕΝ. Σήμερα όμως αναφέρατε πολλά άλλα θέματα. Ποια είναι λοιπόν η πολιτική σας θέση εδώ. Ισχύουν τα όσα είναι γραμμένα στο έγγραφο ή όσα μας είπατε εδώ τώρα, γιατί γεγονό είναι ότι θέλει να κλείσει πολλά θέματα το Κοινοβούλιο πριν από το τέλος ε, της ε, θητείας αυτής. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Πραγματικά, ε, θα απαντήσω λίγο πολύ με τη σειρά που κάνετε τις ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα. Πρέπει να συνηθίσω τον νέο μου ρόλο ακόμα. Προφανώς θα δεχτώ πολλές ερωτήσεις. Κάποιες θα μου απευθύνονται ως ε, Υπουργό Εσωτερικών, κάποιες άλλες υπό τη νέα μου ιδιότητα Κοιτάξτε, προφανώς ε, στο πλαίσιο του Συμβουλίου θα γίνει μια συζήτηση εδώ. Όταν μιλάμε λοιπόν στο ευρωπαϊκό επίπεδο για νομισματικά μέσα και καταλήγουμε σε κάποιες λύσεις για ένα κομμάτι της Ευρώπης, είτε την Ευρωζώνη είτε άλλες χώρες που ακολουθούν άλλες αρχές, πάντα λέμε ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα κράτη εκείνα τα οποία δεν είναι μέλη, στην προκειμένη περίπτωση αυτά που δεν είναι μέλη της Ευρωζώνης. Και νομίζω πως όλοι αντιλαμβανόμαστε τις ε, συζητήσεις και τις αποφάσεις ε, και είναι νομίζω σημαντικό για όλους μας να έχουμε μία συνολική άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβουμε υπόψη όλους όσους ανήκουν σε αυτήν την Ευρωπαϊκή οικογένεια. Η χώρα μας ε, δεν είναι μέλος της Ευρωζώνης και έχουμε κάποια κράτη-μέλη που ακόμα δεν έχουν ενταχθεί αλλά σχεδιάζουν να το κάνουν. Θα ήθελα όμως να πω ότι σε επίπεδο αρχής ε, έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις και αυτή την προσέγγιση θα ακολουθήσουμε στην ε, Προεδρία μας. Θα συζητάμε και θα λαμβάνουμε αποφάσεις για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο για τα μέλη της Ευρωζώνης ή όχι. Όσον αφορά τώρα τον κατάλογο των θεμάτων που θα απασχολήσουν την Προεδρία μας, γεγονό είναι ότι κάποια πράγματα είναι συνεχώς εν εξελίξη. Αλλά το θέμα, όπως είπα, δεν είναι απλά να είμαστε αισιοδοξοί, αλλά να είμαστε αποφασισμένοι. Σας διαβεβαιώ λοιπόν ότι Ε, τα λέω εδώ, θα τα πω αύριο και στο ECOFIN. Θέλουμε να είμαστε ρεαλιστικοί στην προσέγγιση μας. Και να ασκήσουμε θετική πίεση θα έλεγα. Παρά το ότι έχουμε πολύ λίγο χρόνο μπροστά μας, θέλουμε να επιτύχουμε κάποια πρόοδο είμαστε στο τέλος της ε, θητείας, αλλά όπως ως πρόεδρος του ΕΚΟΦΗΝ αυτό θα πω και στο ΕΚΟΦΗΝ και ως υπουργό Οικονομικών ε, της Ρουμανίας θα έλεγα ότι θα είμαστε όσο το δυνατόν πιο αισιόδοξοι με, σε σχέση με τα θέματα αυτά. Mm. Σας ευχαριστώ, Περβάνς Μπερές, για τους σοσιαλδημοκράτες. Κύριε Υπουργέ, μας παρουσιάσατε τις προτεραιότητές σας. Φαίνεται σαν κατάλογος φακέλων που βρίσκεται στο τραπέζι της Ρουμανικής Προεδρίας από όταν άρχισε την προσπάθειά της. Να ρωτήσω σας κάτι. Που είσαστε ο προεδρεύων του ΕΚΟΦΗΝ. Ποια θέματα θεωρείτε ότι πρέπει να προωθήσει η Ρουμανική Προεδρία? Ο κατάλογος των φακέλων που έχετε μπροστά σας τα ξέρω τα θέματα. Εσείς με ενδιαφέρει. Ποια θεωρείτε σημαντικά. Ποια είναι η προτεραιότητά σας. Με καταλαβαίνετε, με ακούτε. Ωραία. Αναφερθήκατε στην επιτευχθήσα πρόοδο τη σχετική με τον επιμερισμό των κινδύνων. Μειώθηκαν οι κίνδυνοι, είπατε. Επί προεδρία σας, η επανεξισορρόπηση πώς θα επιτευχθεί για τον επιμερισμό των κινδύνων. Στους διαδόχους σας θα δώσει το δικό χάρτη που θα έχει εξελιχθεί όσον αφορά τον προπολογισμό της Ευρωζώνης αποτελεί κομμάτι επιμερισμού του κινδύνου αυτό. Αναφερθήκατε στι χώρε που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη. Η Ρουμανία όμως θέλει να προσχωρήσει στο ευρώ. Όπως και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα υπήρχε καθήκον να μεριμνήσετε την ολοκλήρωση της Ευρωζώνης. Διότι για την ώρα δεν μπορεί η Ευρωζώνη να αντιμετωπίσει την επόμενη κρίση, δεν είναι κατάλληλα εξοπλισμένη. Ευχαριστώ πολύ για τα όσα μου είπατε, ερωτήσεις, σχόλια. αυτοί που θα ακολουθήσουν μετά από τη δική μας Προεδρία θα βρουν πράγματα που εξαρτώνται κατά πολύ από τα όσα θα περάσουν το Συμβούλιο εμείς στη δική μας Προεδρία. Εξαρτώνται όμως τα θέματα αυτά και το, από το πώς τα κράτη-μέλη βλέπουν τα διάφορα θέματα. Πώς συνεισφέρουν στη συζήτηση, πόσο έτοιμα είναι τα κράτη-μέλη να συμβιβαστούν στα διάφορα ζητήματα. Υπάρχουν πολλά θέματα προς συζήτηση και μείωση του κινδύνου, η ανακατανομή του κινδύνου είναι ένα από αυτά τα θέματα. Να επαναλάβω ότι κατά την άποψή μου θα προσπαθήσουμε να σημειώσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή πρόοδο. Κυρίως όσον αφορά το πρόγραμμα εργασιών του ΕΚΟΦΗΝ, το θεματολόγιο του ΕΚΟΦΗΝ. Έχουμε ελάχιστο χρόνο, το ξέρω. φτάνουμε στο τέλος της κοινοβουλευτικής θητείας και της θητείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σαν Προεδρία έχουμε καθήκον να υποβάλουμε προτάσεις και να βρούμε συμβιβαστικές λύσεις ούτω ώστε να επιτευχθούν συμφωνίες στα πλαίσια του Συμβουλίου. Όσον αφορά το τεχνικό επίπεδο, στην Κορεπέρ, θέλουμε να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατό στο πλαίσιο της Επιτροπής αυτής. Θέλουμε ισχυρό και ανθεκτικό χρηματοπιστωτικό τομέα. Είναι υποφελές για όλους, για όλα τα κράτη-μέλη. Όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες θέλουν κάτι τέτοιο. Πρέπει να προοδεύσουμε όμως για να το καταφέρουμε αυτό. Ελπίζω να απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις σας, λέει ο κ. Υπουργός, αλλά αν όχι, η κυρία Βέρες. Τα τρία-τέσσερα θέματα θα ήθελα να μου αναφέρετε. Πέρα από τον κατάλογο που παραθέσατε, τα τρία-τέσσερα θέματα που θεωρείτε ότι θέλετε να ολοκληρωθούν αυτά τα θέματα επί Προεδρία σας. Και σαν χώρα που δεν ανοίξει την Ευρωζώνη, τι σημασία δίνεται στα θέματα που σχετίζονται με προπολογισμό της Ευρωζώνης διότι πιστεύω ότι η χώρα σας θέλει να προσχωρήσει το ευρώ. Και τώρα η ευρωζώνη δεν είναι βιώσιμη ως έχει. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Very short. Κοιτάξτε, το Δεκέμβριο του 2018 οι Ευρωπαίοι ηγέτες σε επίπεδο Eurogroup καθόρισαν στόχους. Στόχους που σχετίζονται με δημοσιονομικά εργαλεία σύγκλησης και ανταγωνιστικότητας. Όσον αφορά τώρα την Ευρωζώνη εν γέννη, θα συνεργαστούμε στενά με την ηγεσία του Eurogroup, όπως προανέφερα, ούτω ώστε να υπάρξει σωστό συντονισμό για την αντιμετώπιση των διαφόρων θεμάτων. Έχουμε προθεσμία τον Ιούνιο του 2019. Και μέχρι τότε πρέπει να βρούμε κάποιες λύσεις. Δεν ξέρω αν τώρα μπορώ αμέσως να παρουσιάσω λύσεις όσον αφορά τον προϋπολογισμό της Ευρωζώνης. Δοθέντος ότι η Ρουμανία έχει μια συγκεκριμένη στάση όσον αφορά τη συμμετοχή της Ευρωζώνης συζητήσαμε μια προθεσμία για το 2000, για αργότερα για να μπούμε. Δεν υπάρχει σχετισμός όμως μεταξύ των δύο στόχων. Αναφερθήκατε στον προπολογισμό της Ευρωζώνης. Είναι κάτι ξεχωριστό αυτό. Αυτό είναι ένα θέμα. Και άλλο θέμα η ένταξη της Ρουμανίας στην Ευρωζώνη όσον αφορά τους δικούς μας στόχους. Στην ομιλία μου είπα ότι το Invest EU είναι σημαντικότατο στόχος όπως βλέπω εγώ τα πράγματα, σαν κάποιος που έχει συμμετάσχει σε τέτοιου είδους εργασίες κατά το παρελθόν και ξέρουμε πώς χρησιμοποιούνται αυτά τα μέσα, είναι ένα θέμα σημαντικότατο και ελπίζω να προχωρήσουμε γρήγορα πάνω σε αυτό. Αύριο, όπως είπα, στο ΕΚΟΦΗΝ θα γίνει η πρώτη συζήτηση όσον αφορά αυτό το εργαλείο, αυτό το μέσο. Ήδη υφίσταται μία πρόταση έχει υποβληθεί από τη Ρουμανική Προεδρία. Θα γίνει και άλλη συνεδρίαση το Φεβρουάριο. Και ελπίζω να ληφθεί κάποια απόφαση τότε. Όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο, το ΦΠΑ, σημαντικά θέματα και αυτά. Ειδικοί φόροι κατανάλωση μετά, η βιώσιμη χρηματοδότηση, συμπεριλαμβάνοντα το τριμερή διάλογο. Έχουμε το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο βέβαια. Όπω γνωρίζετε, είναι και αυτό ένα σημαντικό θέμα. Τέλο, όπως έλεγα, το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι σημαντικότατο και θα ακολουθήσουμε παρόμοια προσέγγιση και εκεί. Ούτως ώστε να διεκπαιρεωθεί και αυτό το θέμα. Θέλουμε να ολοκληρώσουμε, να κλείσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα μέτωπα πριν ολοκληρωθεί η πρεδία μα. Ευχαριστώ. Ευπρόσδεκτο αυτό που είπατε για το Invest EU. Να σα υπενθυμίσω εκ νέου ότι είναι κατεπήγον θέμα. Θέλουμε να ολοκληρωθεί ο τριμερής διάλογο. Όσο πιο γρήγορα τόσο καλύτερα. Διότι ο κίνδυνος είναι να μην προλάβουμε και να χάσουμε μεγάλη ευκαιρία. Και η Προεδρία σας να χάσει την ευκαιρία να ολοκληρωθεί ένα τόσο σημαντικό θέμα, σημαντικότατη συνιστόσα, σημαντικότατο εργαλείο για την πρόθεση των επενδύσεων, της απασχόλησης και της ανάπτυξης. Μπεντ Λούκε για το ECR. Θα μιλήσω γερμανικά. Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου. Θα ήθελα να επανέλθω στην απάντηση που δώσατε στον κύριο Μουρεσάν. Από ό,τι κατάλαβα, βασιστήκατε στο ότι όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να ωφελούνται από τα μέτρα τα οποία προβλέπονται στον προεπλογισμό της Ένωσης. Αλλά θα ήθελα να το διευκρινίσετε αυτό. Γιατί οι απαντήσεις σας μέχρι τώρα ήταν γενικόλογες. Θα ήθελα συγκεκριμένα να ρωτήσω για την νομοθετική πρόταση για το Ευρωπαϊκό για την ευρωπαϊκή αυτή λειτουργία σταθεροποίηση ε, Προβλέπει η πρόταση της Κομισιόν πως θα δίδονται άτοκα δάνεια σε κράτη τη Ευρωζώνη και του Μηχανισμού Συναλλαγματικών Ισοτιμιών. Και αυτά θα χρηματοδοτούνται από τον συνολικό προπολογισμό της Ένωσης, δηλαδή από όλα τα κράτη-μέλη. Αλλά δεν θα ωφελούνται όλα από αυτά τα άτοκα δεν μπορούν να ωφελούνται όλα είτε γιατί προσωρινά είτε μονίμως δεν ε, σε μετέχουν είτε στην Ευρωζώνη είτε στον μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η χώρα σας ας πούμε δεν είναι στο μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών αλλά και η Δανία και η Σουηδία δεν είναι μέλη ούτε εκεί ούτε στο ευρώ. Χρηματοδοτούν δηλαδή τα μέτρα αυτά, αλλά δεν έχουν δυνατότητα να ωφεληθούν από αυτά. Κατάλαβα καλά πως αυτό παραβιάζει την αρχή του Συμβουλίου και πως ε, άρα θα απορρίψει το Συμβούλιο την πρόταση της Κομισιόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Ε, μιλάμε εδώ πέρα για την ευρωπαϊκή αυτή, το ευρωπαϊκό μέσο σταθεροποίησης ε, για τις επενδύσεις. Πρόκειται για ένα συγκεκριμένο ζήτημα το οποίο αφορά την ε, Ευρωζώνη. Λοιπόν, όταν μετά μιλάμε για το θέμα του Συμβουλίου και του ΕΚΟΦΗΝ και τις συζητήσεις που θα γίνουν εκεί, Είπατε να διευκρινίσω την απάντηση που έδωσα στον κύριο Μουρεσάν. Είπατε ότι η απάντησή μου ήταν ασαφής. Και με ρωτήσατε, μου ζητήσατε άρα να εκθέσω το σκεπτικό. Λοιπόν, δεν είμαι σίγουρος αν πρέπει να μπορώ να απαντήσω σε όλα αυτά. Αλλά πολλά από αυτά τα ζητήματα σχετίζονται με τα όσα συνέβησαν. Με συγχωρείτε κύριε Υπουργέ, δεν ήταν αυτή η ερώτησή μου για το μέσο. Σας ρώτησα για τις αρχές σας, αυτά τα οποία είπατε στον κύριο Μουρεσάν. Είπατε ότι η αρχή του Συμβουλίου είναι ότι όλα τα κράτη-μέλη θα ωφεληθούν από τα νομοθετικά αυτά μέσα λοιπόν στην συγκεκριμένη αυτή λειτουργία. Θα ισχύσει αυτή η αρχή και άρα θα απορρίψετε την πρόταση της Κομισιόν γιατί κάποια κράτη-μέλη χρηματοδοτούν αλλά δεν ωφελούνται. Ναι. Ε, σας άφησα να διακόψετε λέει ο Πρόεδρος. Ε, δεν θα έπρεπε να γίνει αλλά για να διευκρινίσετε την ερώτηση κύριε Λουκέ. Κοιτάξτε. στην ε, Ρουμανία. Λάβαμε εμείς την απόφαση το 2018 ότι όλα τα κράτη-μέλη ε, θα πρέπει να έχουν ε, μια άποψη η οποία θα είναι σεβαστή και αυτό θα στηρίξουμε. Σας ευχαριστώ. Δεν έχω κάποιον ομιλητή από διάφορες ομάδες. Οπότε περνάμε πάλι στο ΕΛΚ με τον κύριο Φαντερ Κέντελαρ. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω Ολλανδικά. Βάλτε τα ακουστικά σας λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ για την μακρά αυτή εισαγωγή. Έχω δύο ερωτήσεις για κάποια πολύ συγκεκριμένα θέματα και ελπίζω να μπορέσω να πάρω συγκεκριμένες απαιτήσει πρώτα απ' όλα για τις δικαιοδοσίες που δεν συνεργάζονται στον κατάλογο αυτό στον οποίο αναφερθήκατε στην εισαγωγή σας. Είπατε ότι δουλεύετε πάνω σε ένα τέτοιο κατάλογο, ότι θα υπάρξει ενημέρωση για να υπάρχει διαφάνεια στα φορολογικά και ότι θα πρόκειται για έναν κατάλογο που θα έχει κάποιο δυναμισμό, δηλαδή θα αλλάζει. Υπάρχει Σαμό, το Γκουάμα, η Αμερικανική Σαμό, την Πάγκο και τα Virgin Islands για το οποίο θέλω να σας ρωτήσω. Πέντε χώρες που υπάρχουν σε αυτό το κατάλογο. Αυτό τι σημαίνει, ότι οι άλλες δικαιοδοσίες είναι συνεργάσιμες φορολογικά. Υπάρχει περίπτωση πρόσφατα να προσταθούν και άλλες χώρες σε αυτό τον κατάλογο. Ποια είναι η εξολόγηση που γίνεται. Ρωτάω, Ποιε χώρες μπορεί να προσταθούν σε αυτό τον κατάλογο και έχετε σκεφτεί και κυρώσει για αυτές τις δικαιοδοσίε που δεν συνεργάζονται. Δεύτερον, θέλω να σας ρωτήσω για τις ψηφιακές επιχειρήσεις στο ίντερνετ. Είπατε ότι είναι προτεραιότητά σας και αυτό, ότι θέλετε να δουλέψετε όσον αφορά ε, την φορολόγησή του για να παραμένει στο διαδίκτυο. Πώς θα γίνει αυτό λέτε ότι κοντεύουμε να φτάσουμε σε συμφωνία. Έχετε την εντύπωση ότι θα υπάρξει εύκολα μια συμφωνία και συγκεκριμένα πώς γίνεται ο χειρισμός αυτού του φακέλου ώστε το Μάρτιο για παράδειγμα να έχουμε συμφωνία. Ε, ξέρω ότι μάλλον τι θα χρησιμοποιήσετε σαν βάση το γαλλογερμανικό κείμενο ή την αυστριακή πρόταση. Αυτό είναι που σας ρωτάω. Απάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά τη δεύτερη ερώτησή σας και το γαλλογερμανικό κείμενο, η συμφωνία, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν χώρες μέλη που έχουν ήδη πει ότι αν δεν υπάρχει συνένεση, τότε σε ατομική βάση θα ασχοληθούν με αυτήν την συμφωνία μονομερός. Τώρα, εμείς ελπίζουμε ότι θα υπάρξει συζήτηση στο Συμβούλιο και αύριο, για παράδειγμα, στην ημερήσια διάταξη, μεν δεν το έχουμε βάλει, το Φεβρουάριο όμως θα το βάλουμε στην ημερήσια διάταξη για να συζητήσουμε το θέμα της ψηφιακής φορολόγησης και της φορολόγησης των ψηφιακών επιχειρήσεων. Και ελπίζουμε να πετύχουμε κάτι. Θα βασιστούμε στην πρόταση την γαλλογερμανική της προηγούμενης χρονιάς. Οπότε έτσι θα αποφύγουμε διαφοροποιημένη προσέγγιση στα πλαίσια της ενίας αγοράς. Τώρα όσον αφορά τα άλλα ζητήματα, ο, ο ΑΣΕ πολύ σύντομα θα αποφασίσει για μια διεθνή ρύθμιση για αυτά τα θέματα. Βέβαια πρέπει να πάρουμε υπόψη μας και τις συζητήσεις που έγιναν πέρυσι. Είναι ένα περίπλοκο ζήτημα, όπως είπατε κι εσείς. Είναι ένα θέμα όπου οι χώρες μέλη έχουν επιφυλάξεις και γνωρίζουμε πολύ καλά ποιες είναι οι χώρες αυτές οι οποίες δεν είναι πρόθυμες να σπαστούν ε, μια τέτοια ιδέα. Το Φεβρουάριο όμως θα συζητήσουμε στο ΕΚΟΦΗΝ και ελπίζουμε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα συμβασμό ώστε όλες οι χώρες μέλη να εφαρμόζουν τις ίδιες διατάξεις. Για τις δικαιοδοσίες, τις συνεργαζόμενες ημί, το Συμβούλιο εργάζεται πάνω σε αυτό και θα συζητηθεί. Θα βασιστούμε λοιπόν στην ανάλυση που θα γίνει για την κάθε δικαιοδοσία και θα δούμε ποια θα είναι αυτή η ανάλυση. Και ανάλογα θα πράξουμε. Για τον κώδικα δεοντολογίας πρώτα απ' όλα και μετά θα πρέπει να δούμε τι λέει το ΕΚΟΦΗΝ. Δεν μπορώ να σας δώσω τώρα τις λεπτομέρειες, γιατί δεν έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία. Πάντως, όπως καλά γνωρίζετε, είναι μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια ήδη. Και όπως είπα και στην εισαγωγή μου, προσπαθούμε να προχωρήσουμε σε αυτό το φάκελο. Αλλά χρειαζόμαστε περισσότερες ε, λεπτομέρειες για να το πετύχουμε και μόνο τότε θα μπορέσω να σας απαντήσω πλήρως. Σας ευχαριστώ για τους σοσιαλδημοκράτες ο κύριος Φρουντσουλίτσα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Ε, χαρά μας που σας έχουμε εδώ απόψε στην Επιτροπή Οικονομικών θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Οικονομικής Εποπτείας που θα βελτιώσει υποτίθεται τις δυνατότητες που προσφέρονται από την τεχνολογία στον χρηματοπιστωτικό τομέα, τη λεγόμενη FinTech Κάτι πολύ σημαντικό γιατί αφορά ακριβώς τις νέες τεχνολογίες και την ψηφιοποίηση του κόσμου και με δεδομένο το ότι η Ρουμανία έχει θέσει ως στόχο την σύγκληση στην Προεδρία της πρέπει να στηρίξουμε την έρευνα και την ανάπτυξη και την συνδεσιμότητα στην Ευρώπη. Ξέρω λοιπόν πως έχετε συναντηθεί και με τους εισηγητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό και βεβαίως αύριο σας εύχομαι κάθε επιτυχία στην συνεδρία του ΕΚΟΦΗΝ. Θα ήθελα όμως να σας ερωτήσω το εξή. Ποιες είναι οι προτεραιότητες για την Ρουμανία όταν μιλάμε για τον εξυγχρονισμό ακριβώς ε, του μηχανισμού αυτού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Το πακέτο αυτό της ESA ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό για το ECOFIN. Θα μας απασχολήσει στις 12 ε, Φεβρουαρίου, αλλά είναι και αύριο στην ημερήσια διάταξη και στην συνάντηση αυτή θέλουμε όλοι να γνωρίζουν τον στόχο που έχουμε θέσει τελικά και βεβαίω θα μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο, να τροποποιήσουμε ολόκληρο το πακέτο. Αλλά όπως ξέρετε υπάρχουν διαφορετικές απόψεις ε, στο Συμβούλιο. Οπότε θα προσπαθήσουμε ως στρατηγική, ως προσέγγιση αν θέλετε, να προχωρήσουμε αύριο στην συνεδρίαση του ΕΚΟΦΗΝ με τα όσα ήδη έχουν συμφωνηθεί με βάση τη δουλειά που έχει γίνει στο Κοινοβουλίο. Και βεβαίω έχουμε αυτό το πολύ μικρό παράθυρο ευκαιρία για να δούμε τις λεπτομέρειες ε, το, των όσων θεμάτων είναι ακόμα ανοιχτά γιατί βεβαίως έχουν συζητηθεί πολλά ζητήματα στο τεχνικό επίπεδο και στην Κορεπέρ οπότε μετά ελπίζουμε να δούμε αρχές Μαρτίου να γίνουν κάποια πρώτα βήματα στο Συμβούλιο και μετά προφανώς θα επανέλθουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα έχουμε και την πτυχή της ε, καταπολέμησης ξεπλήματος χρήματος μαζί με όλα τα υπόλοιπα θέματα. Όταν μιλάμε λοιπόν για την ενίσχυση της εποπτείας και καταπολέμησης του ξεπλήματος χρήματος κτλ. Γι' αυτό ακριβώς θέλουμε να ενισχύσουμε την πτυχή της ε, σύγκλησης ε, της εποπτείας στα κράτη-μέλη. Αυτό θα έλεγα πως είναι η απάντηση στην ερώτησή σας. Σας ευχαριστώ. Ξανά για το ΕΛΚ. Ο κύριος Μουρεσάν. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Δράτω με τις Δευτέρας ευκαιρίες προς διευκρίνηση σημείων. Ακούσαμε διάφορες ερωτήσεις που παρέμειναν αναπάντητες. Ερωτήσεις κυρίας Μπερές από τους σοσιαλιστές και από τον κύριο Λούκερ. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά την ΟΝΕ. Ναι. Η πρόταση Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Ε, ποια είναι η άποψή σας όσον αφορά τη συμμετοχή χωρών που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη σε αυτό το ταμείο. Τι θα πρέπει να χρηματοδοτείτε. Με ακούτε ή ακούτε το σύμβουλό σας. Τι σύμβουλό σας. Τι είδους χρηματοπιστωτικό, ε, χρηματοδοτικό μηχανισμό θα εξετάζατε. Ποιοι όροι για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και ποιος μηχανισμός χρηματοδοτήσεως τεφίστατο. Η Ρουμανία θα συνέβαλε στη χρηματοδότηση ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου. Αυτά είναι σημαντικά ερωτήματα. Θέλει ο κόσμος να ξέρει τις απαντήσεις. Εδώ συζητούμε αυτά τα θέματα, τα συζητούμε με τους υπουργού που είναι στο πιδάλιο της Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Δεύτερο θέμα προς διευκρίνηση, ελπίζω, από την πλευρά σα. Του φακέλου που θέλετε να προωθήσετε επί Ρουμανική Προεδρία. Αναφερθήκατε στους ειδικού φόρους κατανάλωσης. Στο γραπτό κείμενο τα αναφέρατε. Εδώ είπατε και αναφέρατε άλλα θέματα και μετά μας είπατε βλέπουμε, θα δούμε τι θα γίνει. Όμως οι συνάδελφοί μου θέλουν να ξέρουν ποια θέματα θα διεκπαιρεωθούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου σας. Τρίτον, όσον αφορά τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρώτο εξάμεινο, επί προεδρία σας, το ΕΚΟΦΗΝ θα πρέπει να καθορίσει προτεραιότητες για τον επόμενο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Ποια θα είναι η προτεραιότητα, τρομοκρατία, καταπολέμηση, μετανάστευση, η ασφάλεια των πολιτών, η μείωση τη ανεργία των νέων κλπ. Ποιε προτεραιότητε θα έχετε, διότι η θέση του Συμβουλίου είναι σημαντικότατη σχετικά με τη δουλειά που κάνουμε εμεί στο Κοινοβούλιο για να θέσουμε και εμεί τη στάση μα. Και όσον αφορά και τι διαπραγματεύσει, πώ θα εξελιχθούν, ούτω στο τέλο του έτου να έχουμε τελικά στα χέρια μα ένα προπολογισμό. Σα ευχαριστώ. Απάντηση. Εν συντομία, όσον αφορά τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, θα ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό είναι στην ατζέντα για το ΕΚΟΦΗΝΗ για τις 12 Φεβρουαρίου. Θα το συζητήσουμε το θέμα, θα το αναλύσουμε διόντως και θα κάνουμε την καλύτερη δυνατή πρόταση. Έτσι θα είμαστε θέση να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες ε, του κόσμου. Όσον αφορά το νομισματικό ταμείο που αναφέρατε. Γνωρίζετε άριστα ότι έχει μπλοκαριστεί για ένα χρόνο περίπου το θέμα αυτό. Λυπάμαι, λέει ο κ. Μωρισάν. Εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο ότι επεξεργαζόμαστε το θέμα αυτό. Υπουργό. Σαφή η απαντήση, οι ερωτήσει σα, δώστε τον χρόνο να απαντήσω. Λοιπόν, λέει ο Υπουργό, όπω έλεγα, αυτό το θέμα έχει μπλοκαριστεί στο Συμβούλιο. Και θα ξεκινήσουμε τις συζητήσεις αύριο στο ΕΚΟΦΗΝ και θα δούμε ποια θα είναι η θέση κάθε κράτους μέλους. Έτσι, μετά, θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια διέξοδο. Όπως σας είπα, επί ένα χρόνο έχει αποτελματωθεί το ζήτημα αυτό. Τόσον αφορά τον κατάλογο των θεμάτων. Ήμουν σαφέστατος στην παρουσίασή μου, πιστεύω, την αρχική. Είπα ποιοι είναι οι στόχοι μας, ποιες είναι οι επιθυμίες μας, πώς θέλουμε να συνεργαστούμε με το Ευρωκοινοβούλιο, για να διεκπαιρεώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους φακέλους. Δεν ξέρω αν υπήρξε κάτι που δεν κατανοήσατε εσείς, αλλά εγώ αυτά είπα. Τώρα με ποιον μιλάω εγώ όταν εσείς μιλάτε, αυτό είναι δική μου δουλειά και όχι δική σας. Και ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, είπατε σαφώς ότι για σας η ολοκλήρωση του θέματος Invest EU ήταν κάτι σημαντικό. Σημερίζομαι την άποψή σας, το όραμά σας όσον αφορά τις προτεραιότητες. Πιστεύω ότι είναι καλή προσέγγιση και πρόταση. Κατά κάποιο τρόπο δεν μου είπατε όμως ποιες είναι οι δικές σας προτεραιότητες. Να σας παρουσιάσω εγώ λίστα δικών προτεραιοτήτων και να την εστερνιστείτε. Σας καλώ να την εστερνιστείτε. Αφού τελειώσετε με το InvestEU, Χρειάζεται βιώσιμη χρηματοδότηση. Ταξινόμηση δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί. Οι άλλες πτυχές όμως, οι δείκτες, οι κανόνες περί αποκαλύψεως, περί disclosure, πρέπει να ολοκληρωθεί αυτό. Θα πρέπει το 2 2.2 να διεκπεριωθεί, διότι ξεκίνησε, αλλά είναι σημαντικό πριν το τέλος θητείας να ολοκληρωθεί και επιτρέψτε μου να επιμείνω επί που θα συζητήσετε αύριο στο ΕΚΟΦΗΝ. Και σας έγραψα γι' αυτό μαζί με τον Ότμαρ Καράς, τον συνεισηγητή, η αναθεώρηση των ΕΖΑ. Ξέρω ότι δεν κληρονομείται κάτι εύκολο. Προσέξτε όμως. Μην διαλέγετε τον εύκολο δρόμο της πολιτικής. Ποιος είναι αυτός. Να λέτε υπάρχει ας πούμε ένα συνέστημα όσον αφορά το ξέπλυμα χρήματος. Μας κάνει νέα πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάνω σε αυτό. Λέει, θα αναθέσουμε στην τραπεζική, ένωση, ε, τραπεζική αρχή να το κάνει αυτό. Καλό είναι σαν πρόταση. Αλλά αν δεν αλλάξετε την εξουσία που έχει η τραπεζική αυτή αρχή, επιδεινώνεται η κατάσταση. Την επιδεινώνεται. Δίνεται νέε ευθύνε στην τραπεζική αυτή αρχή, χωρί να δίνετε στην αρχή αυτή τα μέσα για να εφαρμόσει την πολιτική. Λοιπόν, θα πούν η Ευρώπη δεν μπορεί να τα καταφέρει για την καταπολέμηση κατά παρανόμων εσόδων. Και εκεί πρέπει να αλλάξει η διακυβέρνηση της προσπαθίας. Σας ζητά το Κοινοβούλιο να κάνετε ό,τι μπορείτε, ούτω ώστε να υπάρχει μια γενική διαπραγματευτική εντολή. Μετά θα δούμε που θα καταλήξουμε με την πάροδο του χρόνου, που είναι πάρα πολύ λίγος που μας έχει απομείνει. Σα ευχαριστώ. Δεν ήταν ερώτηση ακριβώς αυτό. Ήταν μια συμβουλή την οποία είπατε, θα λάβω υπόψη. Ε, το ερώτημα μου είναι αν συμφωνείτε με αυτές τις προτεραιότητες. Όσον αφορά ε, Όσον αφορά το θεματολόγιο του ΕΚΟΦΗΝ αύριο και το πακέτο ΕΣΑ, μπορούμε να το συζητήσουμε αυτά, όλο το πακέτο σε επίπεδο Συμβουλίου και ξέρω ότι πολλά κράτη-μέλη όσον αφορά το θέμα αυτό δεν συμφωνούν με αυτή την προσέγγιση οπότε θα μπορούσε να κολλήσει το θέμα να δημιουργηθεί ένα διέξοδο και έχουμε μια δεύτερη επιλογή αυτή την οποία συζητήσαμε δηλαδή αύριο να έχουμε πράσινο φως στο Συμβούλιο όσον αφορά το να προχωρήσουμε με μικρά αλλά ασφαλή βήματα και το θέμα για το ξέπλυμα χρήματος να το συζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εναπομένοντα θέματα να συζητούν σε επίπεδο ECOFIN, σαν πακέτο μαζί, από κοινού, αυτά που έχουν μείνει. Αυτό σημαίνει ότι αρχές Μαρτίου περίπου θα είμαστε σε θέση να ασχοληθούμε ολιστικά με το θέμα ECOFIN στο Συμβούλιο. Διαφορετικά δεν θα προλάβουμε. Ίσως αρχές Μαρτίου λοιπόν στο Συμβούλιο να μπορέσουμε να υιοθετήσουμε το υπόλοιπο πακέτο, τα εκκρεμή ζητήματα του πακέτου και η Ρουμανική Προεδρία θα προτείνει κάποιες λύσεις για κάθε στοιχείο, συγκεκριμένες λύσεις που ίσως θα μπορέσουν να τύχουν τις υποστηρίξεις και τις συνενέσεως εντός του ΕΚΟΦΗΝ. Αυτή είναι η δεύτερη επιλογή. Τρίτη επιλογή. Α, όχι. Υπάρχουν μόνο δύο. Δεν υπάρχει τρίτη επιλογή είτε πακέτο συνολικό είτε με βήματα. Και ίσως αυτή είναι ασφαλέτερη επιλογή. Μικρά αλλά ασφαλή βήματα. Πιθανότατα αυτό θα μας δώσει περισσότερες εγγυήσεις για την εξέβρεση λύσεως για τόσο σημαντικό θέμα. Να πω και κάτι ξεκάθαρο όσον αφορά την αυριανή συνεδρίαση του ΕΚΟΦΗΝ. Θα παρίστανται Υπουργοί Οικονομικών, προφανώς. Και βασικός στόχος για το πακέτο αυτό ε, δεν μπορεί να επιτευχθεί εκτός εάν υιοθετηθεί όλο το πακέτο, το γενικότερο, στόχος, μικρά βήματα για την ολοκλήρωση του πακέτου. Όσον αφορά τον κατάλογο των διαφόρων ζητημάτων προς διεκπαιρέωση. Και εδώ πρέπει να πω ότι μου εκφράσατε δική σας άποψη για τα θέματα που είναι σημαντικά. Εγώ ήδη είπα ποια θέματα θέλουμε να προωθήσουμε εμείς σε συζητήσεις του Συμβουλίου και συζητήσει Ευρωκοινοβουλίου και στον τριμερή διάλογο. Νομίζω λοιπόν ότι τα καθόρισα όλα αυτά. Υπήρξε αρκετά σαφή. Μπορώ να τα επαναλάβω αν θέλετε. Αλλά είναι σημαντικό όλοι να σκεφτούν αυτά τα θέματα. Ας Καλησπέρα Υπουργέ και ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ σήμερα το απόγευμα. Θέλω να μάθω ποια είναι η δικιά σας άποψη για την εποπτεία των προπολογισμών των χωρών μελών και τι σημασία δίνετε εσείς στη δημοσιονομική πειθαρχία. Και γιατί το θέτω αυτό. Γιατί πριν από τα Χριστούγεννα η νέα Ιταλική κυβέρνηση πρότεινε έναν προπολογισμό για την Ιταλία με ένα έλλειμμα κάπου στο 2,4% του ΕΠ. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με για να διαπραγματεύσει και τελικά πριν από τα Χριστούγεννα προτάθηκε ένας νέος προϋπολογισμός με 2%. Ε, και δέχτηκε την πρόταση αυτή η Συμβαστικά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αντίθετα, η Γαλλία επίσης έχει δημοσιονομικά μέτρα που φαίνεται ότι θα έχει 3,4% έλλειμμα του χρόνου η Γαλλία με τον προπολογισμό που πρότεινε. Όμως η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου ήταν, πώς να το πω, δεν είπαν τίποτα. Ε, τέλος πάντων δεν ήταν τόσο επικριτική όπως ήταν με την Ιταλία. Και γι' αυτό θέλω να μου πείτε ποια είναι η δικιά σας άποψη από αυτού. Πιστεύετε ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι συνεπή. Πιστεύετε ότι είναι σημαντικό όλες οι χώρες μέλη να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο ή όχι. Ευχαριστώ. Απάντηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Η άποψη εδώ νομίζω ότι είναι σαφής. Οι κανόνες πρέπει να τηρούνται από όλες τις χώρες μέλη. Αυτό αναφέρεται στο σύμφωνο σταθερότητας εξάλλου και αυτή είναι και η δικιά μου άποψη. Και αυτό απαντά και ο πρόεδρος του ΕΚΟΦΗΝ που είμαι εγώ τώρα. Πρόεδρος, ε, ευχαριστούμε. Και η δικιά μας άποψη είναι και ο κύριος Φόξ βεβαίως και γνωρίζει ότι οι κανόνες προβλέπουν ότι το έλλειμμα μετριέται και σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και ε, συγκρίνεται και με την τάση που υπάρχει στον προπολογισμό αν θα αυξηθεί ή όχι και με τις διαρθρωτικές προσπάθειες. Δεν είναι δηλαδή ένα απόλυτο νούμερο, οπότε η κατάσταση ήταν διαφορετική στη μή και στην άλλη περίπτωση. Γίνονται διάφοροι υπολογισμοί, λογιστικοί κτλ. ακριβώς γιατί υπάρχουν ασυμμετρικά μέτρα η διαρθρωτική επιδείνωση στην Ιταλία ε, ήταν πολύ μεγάλη και δίχως προηγουμένου. Δεν μπορούσε να συγκριθεί ούτε καν με τις χειρότερες ερμηνείες που θα μπορούσε να δώσει κανείς για την γαλλική περίπτωση. Δεν κοιτάμε δηλαδή μόνο το νούμερο, το συγκρίνουμε με τα προηγούμενα νούμερα της προηγούμενης χρονιάς. Αν η τάση είναι ανωδική ή όχι. Για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι δηλαδή, έτσι. Δεν είναι όπως ακριβώς το παρουσιάσατε. Δεν εφαρμόζουμε έτσι τους κανόνες. Ωραία. Πολύ χρήσιμη η συζήτηση αυτή. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος συνάδελφος θέλει κάτι να ρωτήσει, ένα κάτσει the αν χρειάζεται. Αλλιώς ολοκληρώνουμε εδώ αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Και ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο του ΕΚΟΦΗΝ που ήρθε εδώ σήμερα. Τον ευχαριστούμε που μας παρουσίασε πολύ συγκεκριμένα το φιλόδοξο πρόγραμμα της Ρουμανικής Προεδρίας. Προσβλέπουμε στη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα κοφήν τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, όχι και πολλούς μήνες, έτσι, γιατί λίγο χρόνο έχουμε μπροστά μας σε αυτό το εξάμεινο που είναι πολύ ιδιαίτερο γιατί είναι ακριβώς μέχρι τις ευρωεκλογές ελπίζω κι εγώ να μπορέσουμε στους λίγους μήνες που μας μένουν να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε όσο γίνεται περισσότερους φακέλους και να τους κλείσουμε. Χρειάζεται βέβαια ιδιαίτερα έντονη συνεργασία μεταξύ μας. Και εμείς να ξέρετε ότι έχουμε κάθε διάθεση για να συνεργαστούμε μαζί σας όσο γίνεται καλύτερα για να πετύχουμε σύγκληση, ανάπτυξη, απασχόληση ε, και συνοχή εδαφική, κοινωνική κλπ. Ωραία, έτσι ολοκληρώνουμε αυτό το σημείο στην Εμερήσια διάταξη και περνάμε στο επόμενο σημείο στην Εμερήσια διάταξη που είναι η απαλλαγή 2017. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Φρουντζουλίτσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. για την συνεδρίαση αυτή. Μάλιστα, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, σκιώδεις εισηγητές για τις ε, παρεμβάσεις τους ε, και την συνεργασία τους για την απαλλαγή των εποπτικών αρχών για το 2018. Τα σχέδια γνωμοδότησης ήταν ούτως ή άλλως αρκετά σύντομα γιατί υπήρχε ο περιορισμός των 1500 ψηφίων και άρα έπρεπε να υποβάλω ο ίδιος πολλές τροπολογίες στο κείμενο. Και γενικώ ε, σε γενικέ γραμμέ ε, τα σχέδια ε, κάνουν κάποιε συστάσει στο ελεγκτικό συνέδριο, σύμφωνα με τι οποίε ε, οι συναλλαγές ε, αλλά και οι πληρωμές και τα έσοδα των λογαριασμών αυτών είναι νόμιμες ε, και τακτικές για να εκπληρώσουν ακριβώς οι αρχές αυτές τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεδομένε και της ανάγκης χρηματοδότηση και τη απόφαση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Βεβαίω θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτό το τελευταίο. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να προβλέψουμε τελικά τι θα γίνει. Επίσης ε, τονίζεται η ανάγκη να διατεθούν περισσότεροι πόροι στην καταπολέμηση του ξεπλήματος χρήματος, να υπάρξει η ενίσχυση της εποπτείας και συνεργασία με διεθνή θεσμικά όργανα ε, εποπτείας των χρηματαγορών. Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή πρέπει να καταλήξει σε κάποια κοινή κατεύθυνση μαζί με την ΕΣΜΑ και την ΕΙΟΠΑ για το πώς ακριβώς θα υπάρξει μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της καταπολέμησης του ξεπλήματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα. Επιπλέον, ε, γίνανε περαιτέρω αναφορέ στην ανάγκη κάποιων προσθήκων στην ΕΟΠΑ σε σχέση με τις αδυναμίες κάποιων κρατών μελών που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη συνεδρίαση όσον αφορά τις αγορές ασφαλιών αυτών των κρατών που κυρίως βρίσκονται στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. δεδομένων και κάποιων ε, αθέμητων πρακτικών κάποιων πολυεθνικών ασφαλιστικών εταιριών. Υπάρχουν κάποιες ε, πολυεθνικές οι οποίες ε, πουλάνε στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη κυρίως και στην νότια, νότιο-δυτική Ευρώπη αν θέλετε, για να είμαι πιο ακριβής ασφαλιστικά προϊόντα χαμηλότερης ποιότητας σε σύγκριση με τα ίδια προϊόντα που πολλούν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με διαφορετικές τιμές. Δεδομένης της ε, φύσης ε, δε της αποστολής της, θα έλεγα πως η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή θα πρέπει να επιδείξει μεγαλύτερη διαφάνεια απέναντι στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, αλλά και στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης αναφέρθηκε και στη συνάντησή μας με τον Ρουμάνο Υπουργό Οικονομικών πως το ανέφερε άλλωστε και η κυρία Μπερές πως η Τραπεζική Αρχή θα πρέπει επίσης να λαμβάνει την κατάλληλη χρηματοδότηση για να εφαρμόζει αυτό το πολύ σημαντικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση του ξεπλήματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Τονίζουμε επίσης ότι θα μειωθούν τα έσοδα της αρχής αυτής με την αποχώρηση του Ενωμένου Βασιλείου και άρα θα ήθελα και πάλι να επισημάνω το τι συνέπειες έχει αυτό και να τονίσω την ανάγκη να βρεθεί επαρκής χρηματοδότηση, να γίνουν κάποιες διευθετήσεις που θα είναι πολύ σημαντικές στο μέλλον το σύστημα το οποίο θα συσταθεί για τη χρηματοδότηση αυτής της αρχής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν όλες αυτές οι αρχές ε, να μπορούν ε, να εκτελούν την έντολή τους με τρόπο συνεπή, ανεξάρτητο και αποτελεσματικό. Και αυτό δεν ε, συνέβαινε πάντα αυτού του λεχθέντος ε, θα ήθελα να πω πως για κάθε σχέδιο απόφασης είχαμε γύρω στις 20 τροπολογίες ε, για τις οποίες είχαμε περίπου 6-7 συμβαστικές προτάσεις σε συνεργασία με τους κοιόδες που κάλυπταν τις περισσότερες τροπολογίες και ήταν μια συγκεκριμένη ενιαία αντιμετώπιση των ε, απαλλαγών των τριών εποπτικών αρχών όσον αφορά τα τεχνικά. Η ψηφοφορία είναι αύριο. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ο κ. Βέρναν Λάγκεν για το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ. Ναι, έχουμε η ιδρύση της αρχές αυτές το 2010 και δεν είναι η πρώτη έκθεση που κάνουμε για τα οργανωτικά τους προβλήματα. Πρόκειται για γνωμοδοτήσεις προς την Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού. Δεν λαμβάνουμε εμείς τις αποφάσεις και ο εισηγητής ε, βεβαίως ε, συνέπηξε τις ε, τροπολογίες σε κάποιες συμβιβαστικές και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω που έλαβε υπόψη τις παρατηρήσεις μας έτσι ώστε η ομάδα του ΕΛΚ μπορεί να υπερψηφίσει τις εκθέσεις χωρίς καμία επιφύλαξη πρώτων. Δεύτερον, αφετηρία για τις εκθέσεις αυτές ήταν οι εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου και εδώ πέρα παρατηρώ μια επιφανειακή αντιμετώπιση εδώ και χρόνια που δεν ε, αναφέρει ούτε τα βασικά προβλήματα όπως παραδείγματος χάρη τα 62 εκατομμύρια ευρώ υποχρεώσεις για το Λονδίνο που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή μέχρι το 2026 γιατί έχει κλείσει τόσο μακροχρόνιο συμβόλαιο ή η ΕΙΟΠΑ e η οποία αναλαμβάνει πράγματα και καθήκοντα τα οποία μεταβίας εμπίπτουν εντός των αρμοδιοτήτων της και επειδή έτσι έχουν τα πράγματα Έχω επισημάνει στο ελεγκτικό συνέδριο τα ζητήματα αυτά και το είδαμε και στην έκθεση της ΑΙΟΠΑ. Τα πράγματα βέβαιω και εκεί πέρα έχουν κάποιες διαφορές. Παραδείγματος χάρη, τη μία έχει αποτελέσματα πολύ ικανοποιητικά, την άλλη επαρκώς ικανοποιητικά. Τι να πω, δηλαδή δεν έχει κάποιο νόημα η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, άμα το πάμε έτσι. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω εδώ πέρα τον εισηγητή για το ότι κατάφερε να κάνει μια χρήσιμη γνωμοδότηση και με βάση και τις τροπολογίες και την βοήθεια των συναδέλφων μπορούμε τελικά να συμφωνήσουμε. Και όπως είπα θα το υπερψηφίσουμε χωρίς κανένα πρόβλημα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Για το ECR, ο Ραφ Πάκετ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τις συμβαστικές. Οι περισσότερες τροπολογίες μας ήταν γνωστές. Ήδη τις είδαμε κάνα δύο φορές τα τελευταία χρόνια. Θέλουμε να διατυπώσουμε ότι το Brexit ενδεχομένως και τονίζουμε ενδεχομένως ότι ίσως συναπάγεται απομάκρυνση από τους στόχους διαστηριότητα που σχετίζονται με πιστώσεις και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα επηρεάσει, εν πάση περιπτώσει, εργασίες και τη λειτουργία των ΕΣΑ. Όλα εξαρτώνται από το κατά πόσο θα υπάρξει Brexit για να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί η ισοδυναμία με τρίτη χώρα μετά τον Brexit. Γι' αυτό θεωρήσα χρήσιμο να προσθέσουμε μια διατύπωση που θα λέει ότι το Brexit, αν χρειαστεί, θα πρέπει να αντικατοπτριστεί στους πόρους περιπροσωπικού και χρημάτων για τα ΕΣΑΣ για να διευκρινίσω κάτι που έθεσαν οι πράσινοι στα σχόλιά τους. Προσδέπω στην αυριανή ψηφοφορία αλλά και σε κάποιες τυχόν διευκρινήσεις για τις αλλαγές που έγιναν. Ευχαριστώ. Για την Άλτε, ο Βολφ Πλίντς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λίγα έχω να προσθέσω. Εγώ είμαι μέλος στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού και εκεί πέρα μας απασχολεί κυρίως το θέμα. Πέρα από το θέμα του ανεπαρκή χρηματοδότηση το θέμα του Brexit που ανέφερε ο εισηγητής. Έχω ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε κάπως πιο ουσιαστικά. Είναι η απόδοση της ε, τραπεζικής αρχής όταν μιλάμε για τα stress test. Δεν τα έκανε πρώτη φορά πέρσι ε, και βλέπουμε ότι κάθε φορά είναι μη ικανοποιητικά. Δηλαδή Έχουμε πολλές και διάφορες τράπεζες που περιγράφονται ως τράπεζες που αποφεύγουν τον κίνδυνο, δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα και μετά από λίγες εβδομάδες ή μήνες ε, βρίσκονται σε πολύ άσχημη θέση. Την τελευταία φορά ε, ήταν το αντίστροφο. Ε, Σορεύτηκαν οι απώλειες των τελευταίων ετών και το συνολικό αποτέλεσμα ήταν χειρότερο σε κάποιες ε, περιπτώσεις. Δεν αντιλαμβάνουμε λοιπόν εάν υπάρχει μια συγκεκριμένη προσέγγιση. Θα πρέπει να υπάρξει κάποια βελτίωση. Την επόμενη φορά που θα γίνουν αυτά ε, θα πρέπει να υπάρχουν ουσιαστικές ε, αλλαγές γιατί ελπίζω πια θα έχουν και διαφορετικές αρμοδιότητες οι εποπτικές αρχές και ελπίζω πραγματικά οι εκθέσεις αυτές να ολοκληρωθούν πριν από το τέλος της εντολής, να συμφωνήσουμε με Κομισιόν και Συμβούλιο και έτσι οι τρεις αυτές υπηρεσίες να έχουν διαφορετικές αρμοδιότητες και στην επόμενη απαλλαγή θα δούμε εάν ο νέος αυτός ρόλος πραγματικά θα είναι ο σωστός. Οπότε αναμένω με ενδιαφέρον το τι πρέπει να γίνει. Αλλά όπως σας είπα, αυτό το οποίο κυρίως ήθελα να τονίσω είναι ότι δεν είναι ικανοποιητικά τα stress test όπως διεξάγονται. Ευχαριστώ. Can Πρόεδρε, μπορείτε να επαναλάβετε αυτό που είπατε, γιατί δεν κατάλαβα ακριβώς. οι δοκιμές αντοχής λέω, που έκανε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ε, για τις τράπεζες. Εκτός μικροφώνου κάποια σχόλια δεν ακούγονται. Πρόεδρος, θα σας δώσω πάλι το λόγο κύριε Σίγητα. Στα πλαίσια του ΚΑΤΣΔΙ μήπως... Εγώ ίσως να πω δύο-τρία πράγματα. Θέλω να πω στον κύριο Κλέντς ότι φυσικά και συμμερίζομαι την ανάλυση του για το τι πρέπει να κάνουμε όσον αφορά τις Ευρωπαϊκές Αρχές Εποπτείας. Εξού και τον καλό με τον ίδιο τρόπο να προσπαθήσει να πείσει την κυβέρνησή του για τη θέση που θα υιοθετήσει αύριο στο ΕΚΟΦΗΝ. Γιατί αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας, ή ένα τέλος πάντων από τα κλειδιά της επιτυχίας, για να υπάρχει ενιαία εντολή για τις εποπτικές αρχές. Και το ξέρετε οι δυνατότητες να επηρεάσω εγώ την κυβέρνησή μου είναι να λέει ο κύριο Κλίντ. Η κυρία Μπέρε, εντάξει, καταλαβαίνω. Πάντως, συμφωνώ μαζί σας να έχουμε ευρία εντολή. Τώρα, όσον αφορά αυτά που είπε ο εισηγητή για τι συμβάσει ασφάλισης, έχετε δίκιο που επιμένετε για τις συμβάσεις αυτές, γιατί πρόκειται για τις δημοσιονομικές αγορές, έτσι, οπότε χρειάζεται μια διασφάλιση η ευαισθησία στα διασυνοριακά θέματα είναι μεγάλη. Ξέρετε, υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις ασφαλιστικές που μπορεί να έχουν δύο διαφορετικά στάνταρτ για τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Η διανομή δηλαδή των προϊόντων ασφάλισης μπορεί να είναι διαφορετική από χώρα σε χώρα. Και αυτό είναι πολύ ευαίσθητο Ε, σε μερικές περιπτώσεις, μάλιστα, ε, μια ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να έχει απλώς μια επιχείρηση θηρίδα σε κάποια χώρα και να μην αντιστοιχεί αυτό καθόλου στα επίπεδα εγγύησης που θα περίμενε κανείς από ασφαλιστικές εταιρείες. Είναι πράγματα που με τον κύριο Κλίντς προσπαθήσαμε να διορθώσουμε στην ε, περίπτωση της ΙΟΠΑ προκειμένου να υπάρχει ένας καλύτερος συντονισμός. Πάντως, αυτό που μπορούμε να πούμε για την απαλλαγή σας, ό,τι μπορούμε να πούμε δηλαδή από αυτά που λέτε, ευχαριστώ. Αυτά είχα να προσθέσω κι εγώ και τώρα σε εσά ο λόγος για να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα. Α, μια στιγμή, μια στιγμή. Παρακαλώ. Ναι, μια σύντομη παρατήρηση υπερβάνσου. Ο έλεγχος ε, του προπολογισμού υπάρχει για να ελέγχουμε εάν οι δαπάνες έγιναν αποτελεσματικά και με τρόπο νόμο. Τώρα, αν είναι να μπούμε σε ουσιαστική συζήτηση, αντιλαμβάνομαι και την δική σου την παρατήρηση και του συναδέλφου, πρέπει να γίνει μια γενικότερη συζήτηση, αλλά πέρα από τα αντικειμενικά γεγονότα που μας απασχολούν εδώ πέρα και τα όσα λέει το ελεγκτικό συνέδριο. Δηλαδή, σωστή η συζήτηση αυτή, αλλά δεν είναι η κατάλληλη ώρα. Αυτό ήθελα να πω εγώ μόνο. Εν αυτή περίπτωση δεν ξέρω ακριβώς, συνάδελφε, ποια ήταν η έννοια της παρεμβάσεώς σας όσον αφορά τις εργασίες του ελεκτικού συνεδρίου. Υπάρχει προς συζήτηση. ενδελεχή συζήτηση, διότι παρατηρώ ότι εντολή για το ελεκτικό συνέδριο είναι εξέταση των διαφόρων ε, λογιστικών στοιχείων. Έχουμε ένα θεσμό που αναλύει τις επιδόσεις των πολιτικών που δεν είναι στην εντολή του. Νομίζω ότι αυτό είναι το πνεύμα της παρέμβασής σας. Με τα χαρά σε αυτό το συζητήσουμε δελεχέστερα. Κύριε Σιγητά, έχετε το λόγο για να ολοκληρωθεί το θέμα των λογαριασμών στα πλαίσια της απαλλαγή, που δεν απαγορεύει βέβαια να αναφέρεται και κάποιο άλλο πολιτική σημασία θέμα. Όταν το καλεί επικαιρότης. Κύριε Σιγητά, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Για μία ακόμη φορά θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ε, σκιώδης Να υπογραμμίσω πρέπει ότι όλες οι συστάσεις και όλες οι τροπολογίες που υπευλήθησαν εισήχθησαν στις συμβαστικές τροπολογίες στις οποίες καταλήξαμε. Όλες ταυτόχρονα. Βλέπω ότι γίνονται συζητήσεις όσον αφορά την εποπτεία των εθνικών αρχών. Αρκετά σημαντικό θέμα. Να αυξηθεί αυτή η εποπτεία. Για μία ακόμη φορά να υπογραμμίσω ότι είναι σημαντικό ότι θέλουμε να πετύχουμε σύγκληση μέσω, αυτό, μέσω αυτών που προτείνουμε. Σύγκληση των εποπτικών μηχανισμών σε όλα τα κράτη-μέλη. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοια σύγκληση των διαφορών εποπτικών μηχανισμών σε όλα τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές, αν κάνουμε μια ανάλυση της καταστάσεως. Ελπίζουμε, βέβαια, ότι με τη νέα Προεδρία του Συμβουλίου, όπως μας είπε ο Ρουμάνος Υπουργός Οικονομικών της, το ΕΚΟΦΗΝ, θα πραγματοποιηθεί σύγκληση των εποπτικών μηχανισμών όσον αφορά το ελεκτικό συνέδριο. Συνεχώς ακούω τα ίδια. Τελικά το ελεκτικό συνέδριο, αγαπητοί συνάδελφε, πρέπει να πει ένα πράγμα αρκετά σημαντικό για τα τρία θεσμικά όργανα, τα υποπτικά. Ότι οι λογαριασμοί είναι νόμιμοι, και πρέπει να τοποθετηθεί επί της νομιμότητας και του τακτικού χαρακτήρα, του κανονικού χαρακτήρα των λογαριασμών. Αυτό υποχρεούται να κάνει το ελεκτικό συνέδριο. Ευχαριστώ. Ελπίζω αύριο να ψηφίσετε την απαλλαγή. Ευχαριστώ. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των παρεμβάσεων που ακούστηκαν, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η ψηφοφορία θα είναι εύκολη αύριο. Αυτά τα τρία θέματα της απαλλαγής θα ψηφιστούν στη συνεδρίασή μας την αυριανή. Οπότε ολοκληρώσαμε την ημερήσια διάταξή μας. Θα ξαναρχίσουμε τις εργασίες μας αύριο στις 9, μια κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Περιβάλλοντος για να εξετάσουμε τις διάφορες τροπολογίες για το θέμα αυτό της ε, ταξινόμησης των προτεραιοτήτων. Ευχαριστώ.